Good morning. We are going to do uh, Καλημέρα. Θα κάνουμε ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία με την ηλεκτρονική μας κάρτα. We are going to proof. The first is going to be just a proof. Θα κάνουμε μια δοκιμή αρχικά για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Βάλτε σας παρακαλώ τις κάρτες σας και ψηφίστε ό,τι θέλετε como veis, aquí veis cuántas tarjetas hay. we are just doing a test to vote. Δοκιμή κάνουμε. We are 28 persons inside and now 18 people vote. Είμαστε 28-18 έχουν ψηφίσει. Ψηφίστε σα παρακαλώ, απλά για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Okay. Okay, so... Ωραία. Θα μιλήσω ισπανικά. Διότι ε, μιλάω πιο γρήγορα στα ισπανικά. Καλημέρα σας λοιπόν θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία πάνω στην, ετήσια έκθεση, πάνω στην έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή κατά το 2018. Και ξεκινάμε με την τροπολογία 22. Έναξη της ψηφοφορίας λήξη. Ψηφίσατε μάλλον όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 άρχεται η ψηφοφορία. 23 και 24 μαζί. Πιθάμος αβοταθείων. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα. Συμβιβαστική. Υπαριθμών 2. Ψηφίζουμε. Αδοπτάδα. Γκρίνεται. Και. 27. 27 παράγραφος 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτωτα. 26, 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Ψηφίζουμε. Σε τα Πέρας. Απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στο 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του κυρίου Βίντε. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 34. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Ψηφίζουμε. Σε Πέρας. Συμβιβαστική. 3. Ψηφίζουμε. Βάλε. Σε Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβιβαστική 3β. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα στην συμβαστική τέσσερα ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται ομόφωνα αλλά ψήφισε ένας παραπάνω από το Renew. Άρα θα πρέπει να δηλώσει αποχή κάποιος από το Renew. Ε, γιατί έχουμε εδώ όλου τα τακτικά μέλη και κάποιον πληρωτεί. Άρα συνεχίζουμε, αλλά κάποιος θα πρέπει να μην ψηφίσει από το Ρινιού τώρα. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. τέσσερα. 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Σαράντα Σε τρία τμήματα είναι, οπότε πάμε στο πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 49, τμήμα 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 49, τμήμα 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 50. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. 50 το 2. Ψηφίζουμε. Πέρας και απορρίπτεται. 51 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Β. Επομένως. Και αρχίζει την ψηφοφορία τώρα. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Και πάλι ψήφισε ένας παραπάνω από το Ρήνιο. Όχι, τι γίνεται. Δεν ξέρω, έτσι λέει το μηχάνημα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα ψηφορίας. Και τώρα πάμε στο 55-1. 55-1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 55-2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 56. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 57. Ψηφίζουμε. Σε θύρα Πέρας. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. 58. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Ψηφίζουμε. εγκρίνεται και πάμε στο 61 ψηφίζουμε πέρας και απορρίπτεται 62 ψηφίζουμε εγκρίνεται 63 ψηφίζουμε κύβο Πέρας. Απορρίπτεται. 64. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 66. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 67 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 68 ψηφίζουμε. Πέρασε. 69 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 70 ψηφίζουμε το 2. 70 το τμήμα 2 ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 70. 71. διορθώνει η πρόεδρος. Το 71. 71 Γεωργούλη. Ψηφίζουμε το 71. Κατέπεσε. Οπότε δεν γίνεται ψηφορία για το 71. Κατέπεσε. Και πάμε στην συμβιβαστική 9. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στο 74. Ψηφίζουμε το 74. Πέρας. Εγκρίνεται. 75. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται και πάμε στο 76 τμήμα υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 76 τμήμα 2. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 77. Ναι, 77. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 78 ψηφίζουμε. Σε θύρα βουτά. Πέρας. Εγκρίνεται. 79 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 80 ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 81 Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 82. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται 84. Πέρας. Εγκρίνεται. 85. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 86. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 87. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του Κριστιαν Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να προσθέσουμε τη λέξη aviation, αερομεταφορές, μετά το European. Με άλλα λόγια, η ε, τροπολογία θα λέει ε, επικροτή ε, τα, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αερομεταφορών. Ωραία, τέλεια. Οπότε, Ψηφίζουμε το 88 του κυρίου Τέρχες. Ψηφίζουμε. Προφορική τροπολογία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Πέρας το, το 89. Πέρας. Εγκρίνεται. 90. Πέρας. Εγκρίνεται. 91. Πέρας. Εγκρίνεται 92. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται 93. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 94. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 95. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 96. Πέρας. Εγκρίνεται. 97. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. 98, Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 2. Σιωτιολογικέ παραγράφου. Ψηφίζουμε το 2. Πέρα. Απορρίπτεται. 3. Ψηφίζουμε. Πέρα. Απορρίπτεται. 4. Ψηφίζουμε. Πέρα. Και 5. Ψηφίζεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έξι ψηφίζουν. Πέρας. Εγκρίνεται. Επτά. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. Οκτώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Εννέα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εκρίνεται. 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 1. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 15. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 16. εγκρίνεται 17 εγκρίνεται 18 ψηφίζουμε πέρασε εγκρίνεται 19 ψηφίζουμε πέρασε εγκρίνεται 20 ψηφίζουμε πέρασε Εγκρίνεται. 21. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, παράγραφοι αιτιολογικές ε, υπαριθμών 1 τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και απορρίπτεται το 1. Και τότε το σύνολο του κειμένου ψηφίζουμε ahora. Se cierra votación. A ah, ver, todo el mundo. Falta. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Κάποιο δεν έχει ψηφίσει. Πέρασε ο φορέα. Η 28 προς ένα με μία εποχή. Συγχαρητήρια. Και ευχαριστώ πολύ. Okay. Let's continue. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Και όποιο θέλει να αποχωρήσει από την αίθουσα, ας το κάνει γρήγορα, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε με τις συνεδρίες τη Επιτροπής μας. Με ακούτε, σας παρακαλώ. Okay, I'm going to speak in Spanish. Θα μιλήσω ισπανικά. al τώρα προχωρούμε στο σημείο 17 της ημερησίας διάταξης Πρόκειται για μια δημοσία ακρόαση όσον αφορά το ΦΑΤΚΑ και επίσης τις εξοεδαφικές της επιπτώσεις για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγάλη μας ε, χαρά θα κάνουμε αυτή την ε, ακρόαση που την έχει οργανώσει η Επιτροπή μας. Επίσης καλωσόρισαν οι συνάδελφοι από τις Επιτροπές ε, ΕΚΟΝ και ΛΥΜΠΕ. Τους ευχαριστούμε για όσα έκαναν για το θέμα μέχρι σήμερα και επίσης ε, περιμένουμε την συμμετοχή σας στην συζήτησή μας και πρώτα-πρώτα ε, καλώς όρισε ο Αναφέρον και θα του δώσουμε το λόγο για μια πρώτη παρέμβαση δεκάλεπτη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξεκινάω αμέσω με την αναφορά μου. Την εισαγωγή μου, δηλαδή. Ε, πολλά νέα πρόσωπα και πολλά οικία πρόσωπα, οπότε θα έλεγα να σας δώσω ένα ιστορικό της αναφοράς μου που έχει ε, ένα παρελθόν πενταετές σχεδόν μια γενική επισκόπηση του τι συνέβη και τι δεν συνέβη. Όσον αφορά την απάντηση που έχω λάβει από τα θεσμικά όργανα, 1 Σεπτεμβρίου του 2016 υπέβαλα την αναφορά πριν από το GDPR και ένα από τα βασικά ζητήματα που ασχολεί, με τα οποία ασχολείται η, η αναφορά μου είναι το πώς ο ΦΑΤΚΑ παραβιάζει τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δοκιμάτων. Και ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτω εγώ στην αναφορά μου είναι το ζήτημα της αναλογικότητας. Δεν θα, τα, ε, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, απλά αυτή η μαζική μεταφορά δεδομένων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σχετικά με Ευρωπαίους πολίτες προς, την, ε, προς τις θεωρώ ότι δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας και πιθανότατα παραβιάζει και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. νομοθεσία. Πόσο μάλλον όλα αυτά συζητούνταν πριν από το GDPR. Από το 2016 λοιπόν προσπαθώ να λάβω απαντήσεις από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ε, Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ε, Προσωπικών Δεδομένων. Email, επιστολές έχω στείλει άπειρε άπειρες ε, από το 16 και με αγνοούν. Προσπάθησα μάλιστα ε, να απευθυνθώ και στον διαμεσολαβητή, ε, προκειμένου να ε, επιταχυνθούν οι διαδικασίες και στις 8 Φεβρουαρίου του 2019 επιτέλους μου απάντησε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29, τρία χρόνια αργότερα δηλαδή, και αυτή η απάντηση στην πραγματικότητα απέφευγε το, το, το ζήτημα, προσπαθούσε δια, της διολίστησης να, ε, να μην απαντήσει και χάρη στην Επιτροπή του, Πέτη και την ε, δουλειά που ε, έχει κάνει το Κοινοβούλιο, ο καθηγητής Γκαρμπαρίνο ε, απέστειλε μια έκθεση στην Επιτροπή σας, όπου επισημαίνει τις διάφορες παραβιάσεις του GDPR. Πάλι προσπάθησα να απευθυνθώ στον Ευρωπαίο Επόπτη με email, με επιστολές και το 2019 η απάντηση που έλαβα είναι ότι το ΦΑΤΚΑ είναι μια διαδικασία σε εξήλιξη και δεν έχουμε λάβει κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Ούτε μπορούμε να σας δώσουμε σχόλιο αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πότε θα ληφθεί απόφαση. Αυτά όσον αφορά τις αρχές προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι θεμελιώδες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών Δυστυχώς ε, δεν ξέρω αν έχει ε, προκύψει κάτι στο μεσοδιάστημα. Ελπίζω σήμερα να λάβουμε, κάτι, ε, να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες. Υπήρξε και ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου το 18, όπου το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Πόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να εξετάσουν το θέμα. Άλλα εκτελεστικά όργανα και η Κομισιόν συγκεκριμένα έχουν συμμετάσχει, η συγκεκριμένα η Κομισιόν έχει συμμετάσχει σε όλες τις ε, ακροάσεις που έχουν γίνει ε, εδώ στην ΠΕΤΗ. Στην πραγματικότητα όμως ε, αποφεύγει αυτό το θέμα, δεν απαντά ποτέ, στέλνει χαμηλόβαθμους αξιωματούχους στις επιτροπές μας, χρησιμοποιεί έολα επιχειρήματα, αποφεύγοντας να, να δει τα ζητήματα αυτά κατάματα. 25 άνθρωποι από την, ε, έχουν έρθει σήμερα εδώ μαζί μας, κατά τύχη ε, Αμερικανοί, έχουν έρθει από όλη την Ευρώπη, από τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ίσω και άλλε χώρε. Είναι ζήτημα πραγματικό. Είναι υπαρκτοί άνθρωποι και μάλιστα έχουν, έχουν έρθει εδώ στην επιτροπή σα σήμερα οι άνθρωποι αυτοί. Η Κομισιόν το αγνοεί το ζήτημα, του περιφρονεί αυτού του ανθρώπου. Έχουμε κάποιε ιδέε, κάποιε ε, υποψίε γιατί τηρεί αυτή τη στάση η Κομισιόν. Προφανώς έχει να κάνει με πολιτικό κόστος και πολιτικό όφελος. Ίσως θα μπορούσε να είναι ότι ο φόβος ότι αν ε, καταπολεμήσει το ΦΑΤΚΑ, καταπολεμάς ταυτόχρονα και το CRS, αυτό αυτή την κοινή βάση δεδομένων που μας βοηθά να καταπολεμήσουμε το διεθνές οικονομικό έγκλημα. Γεγονός πάντως είναι ότι δεν γίνεται να αγνοούνται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών των δεδομένων για λόγους πολιτικού ωφέλους. Εγώ θα μιλήσω ανοιχτά. Έρχομαι εδώ και τέσσερα χρόνια στην Επιτροπή σας και ε, δεν έχει γίνει τίποτα. Πρόκειται για μια στάση μειοπική, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τους, ε, το, τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και δεν ασχολείται καν με το γεγονός ότι παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εγώ είμαι φιλοευρωπαίος, είμαι μισό Ιρλανδός, μισός Γάλλος. Κάθε Σάββατο παίρνω τα παιδιά μου και ε, τα περνάω και περνάμε μέσα από τον, ε, την λεωφόρο Ζαν Μονέ. Ο Ζαν Μονέ που από το 75 έως το 75 συνέβαλε στην οικοδόμηση αυτού του ε, ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Εγώ λοιπόν ως πεπισμένος φιλοευρωπαίος πολίτης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μας ακούει τουλάχιστον γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μην ακούει εμένα αλλά νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να κάνει διάφορα πράγματα, από τα οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν διερεύνησε το ζήτημα δεν, που σχετίζεται με την ΦΑΤΚΑ. Δεν μας μιλάει. Δεν έχει κάνει τίποτα. Και μάλλον θα, έρθει εδώ, θα, έρθει, θα έχει έρθει εδώ και θα μας πει ότι είναι ζήτημα αμερικανικό, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Υποθέτω. Κάτι πιο θετικό να κλείσω. Τι μπορεί να γίνει όταν η εκτελεστική εξουσία ξυπνά και κάνει κάτι. Έχουμε και κάποια πρόσφατα παραδείγματα. Λάβαμε πολύ συγκεκριμένη ε, ισχυρή ε, δράση ε, στην, ε, ε, ελήφθη μάλλον στην, στη Γαλλία όπου πέρασε ένα ψήφισμα και αποδεικνύει το ψήφισμα αυτό ότι μπορούν να γίνουν πράγματα το Μίνο Σνέλ στην Ολλανδία, ο, ο Υπουργός μάλλον βιομηχανία. τι έγινε, πήγε στην Αμερική και πολύ γρήγορα οι Αμερικανοί ε, αναγνώρισαν ότι είναι πρόβλημα και αναγνώρισαν και μια μερική αμνηστία σε Αμερικανούς πολίτες που έχουν διπλή υπηκότητα. Δεν ήταν ιδανική λύση, αλλά ήταν κάτι. Βλέπουμε ότι οι εγχώροι πολιτικοί ξυπνάνε. Αλλά δυστυχώς καλέσαμε και την Υπουργό ε, βιομηχανία των ΗΠΑ που ε, δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα μαζί μας. Όμως ε, υπάρχουν τέλος πάντων πολλοί πολιτικοί οι οποίοι είναι υπέρ του να προστατευτούν τα, τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και με αυτό θέλω να, να κλείσω. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τη διάκριση των εξουσιών. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Όργανο, το οποίο μα υποστηρίζει εδώ και τέσσερα χρόνια. Βλέπω την Τζου, τη Σόφη, όλου αυτού του ανθρώπου που μα έχουν ε, βοηθήσει σημαντικά. Και σα ευχαριστώ θερμότατα εσά ω νομοθέτε. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Εξουσία, η οποία μα αγνοεί και εμεί οι πολίτε τι, τι, τι καλούμαστε να κάνουμε για να, να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τη διάκριση των εξουσιών. Αυτό που μας λέει η διάκριση των εξουσιών είναι ότι όταν η εκτελεστική εξουσία μας αγνοεί μπορούμε να στραφούμε στη δικαστική εξουσία. Και γι' αυτό χαίρομαι που βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι εδώ, γιατί εκείνοι γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει όταν παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κάτι που συμβαίνει με το ΦΑΤΚΑ. Οπότε θα στραφούμε κατά πάσα πιθανότητα στη δικαστική εξουσία, αφού η εκτελεστική μας αγνοεί, γιατί ε, σε αυτήν τουλάχιστον μπορούμε να βασιστούμε μαζί βεβαίω και με την νομοθετική εξουσία τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά εισαγωγικά και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα με μεγάλη μου χαρά να σα παρουσιάσω το πρώτο πάνελ όσον αφορά τι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε. Ε, έχουμε τώρα το, τους εξή. Πρώτα-πρώτα τον κύριο Σεν ε, Μαρτέν, στην συνέχεια τον κύριο Ράιερ Γιάνσεν, ο οποίο προέρχεται από τι ε, κάτω χώρε και είναι υποδιευθυντής ε, του Υπουργείου Οικονομικών και επίση ο Ρότζερ Κάιζερ ε, από την ε, Τραπεζική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ε, για 10 λεπτά έχετε το λόγο κύριε Σέμαρτα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μας ανατέθηκε σε μένα και στον κύριο Μάρκ Λεφύρ, τον ε, βουλευτή, εδώ και 1,5 χρόνο, να δούμε τι γίνεται με αυτό τον Accidental American το πρόβλημα αυτό. Πρόκειται για ένα θέμα, για μια έρευνα που αφορά αυτήν την ε, επίγουσα ε, προβληματική που αφορά την Γαλλία. Δηλαδή το τι γίνεται με αυτές τις δυσμενείς διακρίσεις σε επίπεδο τραπεζικό. Αυτά τα λέω προσαγωγικά για να καταλάβετε πώς ε, σήμερα ασχολούνται με αυτό το ζήτημα οι βουλευτές και υπάρχει και μια αρνητική πλευρά. Είναι το θέμα της ΦΑΤΚΑ, του ΦΑΤΚΑ, που αφορά αυτή την εξοεδαφικότητα σε σχέση με το Αμερικανικό δίκαιο. Ε, γι' αυτό λοιπόν ασχοληθήκαμε και πάρα πολλοί μας, ε, το υπέδειξαν. Ε, εγώ προέρχομαι από την περιφέρεια του Παρισιού ως βουλευτής, άλλοι το έχουν επισημάνει που έρχονται από τη Βρετανία, αλλά τέλος πάντων αφορά όλη τη Γαλλία αυτό το θέμα και αφορά και αυτούς που έχουν διπλή ηθαγένεια, γαλλική και αμερικανική. Ε, και οι δύο λοιπόν, και εγώ και ο συνάδελφο, συμμετέχουμε στην Οικονομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου εδώ και ένα μισή χρόνο. Εργαστήκαμε για αυτό το θέμα και τελικά τον Μάιο του 19 καταλήξαμε σε μια έκθεση. Ε, σοκάναμε, είδαμε όλους εμπλεκόμενου για αυτή τη μελέτη μας, την έκθεσή μας και είδαμε και ε, αυτούς τους ε, πολίτες, τους Occidental Americans που έχουν το δικό τους φορέα αλλά επίσης ε, ε, συναντήσαμε πολλούς και από την γαλλική διοίκηση και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε βεβαίως επίσης συναντήσαμε τον Πιέρ Λελούς, παλαιό βουλευτή, Φρεντερικ Λεφεύρ και αυτός παλιός βουλευτής που είχε ασχοληθεί με αυτή την εξοεδαφικότητα και το δίκαιο. Και ήρθαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, επί Μπερές και Ροζιέ και επίσης συναντήσαμε διάφορους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επισκεφτήκαμε την Τελωνική Διεύθυνση, Οικονομικές Υπηρεσίες, την Ένωση Αγορών και Κεφαλαίων και άλλες ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν γινόταν αυτή η ακρόση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφήγη το ζήτημα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε κάποια σχετική εντολή από τα κράτη-μέλη. Ε, οπότε τα πράγματα δεν δίρκεσαν και πολύ ε, γιατί η έκπληξή μας ε, έπρεπε να έχει ρητός προβλεφθεί. Μίλησαμε φυσικά και με την Τραπεζική Ένωση, από την οποία προέρχεται ο κύριος Κάιζερ και επίσης συναντήσαμε και εκπροσώπους ε, της ε, ε Αμερικανικής Κυβέρνησης, φυσικά την Εφορία, ε, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και στην Ουάσιγκτον μιλήσαμε ένα σωρό βουλευτές και ε, γερουσιαστές. Όλοι ε, πήραν πολύ σοβαρά το ζήτημα γιατί ακριβώς έχουμε εκτός από τους ε, Γάλλους και τους Αμερικανούς που ζουν στην Γαλλία τους εκπατρισμένους και αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και ελπίζουμε ότι θα πιάσει τόπο η δουλειά μας. Οπότε ακριβώ έγινε έρευνα, ε, μαζέψαμε πληροφορίες στην Αμερική. Δεν θα σας πω όλο το νομικό πλαίσιο που άλλωστε το γνωρίζετε, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε ε, κάποιους με διπλή ηθαγένεια, που τυχαία ή από μια σειρά συμπτώσεων πήραν την Αμερικανική ηθαγένεια. Ε, δεν αφορά όλους όμως με την διπλή ηθαγένεια. Αφορά το θέμα τους Γάλλους ή και άλλους που έχουν και την Αμερικανική ε, ηθαγένεια από τους γονείς τους, αλλά ποτέ, ποτέ ε, δεν έχουν καλυφθεί από κάποιες κρατικές υπηρεσίες ε, παρά τις σχέσεις τους με τις παρά βέβαια ε, το ότι προβλέπει σχετικά το Σύνταγμα. Ε, Επομένως, αν κάποιος έχει την Αμερικανική ηθαγένεια με το use σόλι, τότε de facto κανείς έχει ε, φορολογικές υποχρεώσεις, εξού και η ΦΑΤΚΑ, όπως και τα γνωρίζετε. Οπότε η διορθυμία στη Γαλλία, αυτό ήταν το ζήτημα, είναι ότι γιατί τελικά έχουμε περισσότερους τέτοιους ε, ανθρώπους στη Γαλλία και όχι αλλού. Να δούμε τι θα πει ο συνάδελφος από την Ολλανδία. Ίσως έχουμε πιο πολλούς στη Γαλλία με διπλή ηθαγένεια τέτοιες περιπτώσεις γιατί ε, έχουν σχετική πολιτική οι γαλλικές τράπεζες. Αυτό υποθέσαμε. Δεν λεπτά έχω ποτέ να σα τα πω πάρα πολύ γρήγορα για τι συγκεκριμένε μου προτάσει. Αλλά το θέμα είναι γιατί αυτοί οι Γαλλοαμερικανοί, όλοι αυτοί επομένω, θεώρηθηκαν ότι φύσατε δημιουργημένη διάκριση από τι γαλλικέ τράπεζε και δεν μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό στην τράπεζα. Πολύ συγκεκριμένο αυτό. Έχουν πρόβλημα επίση για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ε, Κάποιο δεν μπορεί να κάνει δηλαδή κάποια ασφάλιση ζωή, δεν μπορεί να κάνει ε, να πάρει στεγαστικό δάνειο, προβλήματα καθημερινά δηλαδή. Και θεωρούμε ότι αυτό αφορά κάποιες μεγάλες τράπεζες, κάποιους ομίλους τραπεζικού στη Γαλλία. Σχετίζονται με τη ΣΥΠΑ σε επίπεδο εμπορικό, ε, κάνουν συναλλαγές σε δολάρια και βέβαια συμμορφώνονται με την Αμερικανική νομοθεσία. Πάντως υπάρχει η σχετική διακυβερνητική συμφωνία, ότι δηλαδή έτσι καταλήγουμε σε αυτή τη δυσμενή διάκριση με την εφαρμογή Αμερικανικής νομοθεσίας από τις γαλλικές τράπεζες. Άρα θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια λύση, ε, αν όχι σε εθνικό επίπεδο, ελπίζω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρία λεπτά και μου μείνανε και να σας πω τις προτάσεις μας. Πρώτα πρώτα, είπαμε θα πρέπει να γίνει συνεννόηση πανευρωπαϊκή. Να γίνει κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Αλλά πρέπει να δούμε θα πρέπει, μπορεί να γίνει από Γαλλίας, αλλά και είπα. Θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα από το ΕΚΟΦΗΝ, το είπαμε αυτό από τον Μάιο. Από τότε υπήρξε μια ομάδα υψηλού επίπεδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 28 Οκτωβρίου εξετάστηκε το θέμα. Θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει με τον κανονισμό 2271 του 91 όσον αφορά τους λογαριασμούς και τον νόμο ΦΑΤΚΑ διαπραγματεύσεις επομένως με τις εμπλεκόμενες χώρες. Να αναθεωρηθούν τα κατόφλια όσον αφορά το πότε θα πρέπει να γίνεται η διαβίωση των σχετικών ε, πληροφοριών και των ε, δηλώσεων στα πλαίσια της συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και φοροδιαφυγής. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός ε, του ΦΑΤΚΑ. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι κατόφλι θα έχει αυτός ο νόμος για να μην φύγονται πολλοί συμπολίτε μας. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί ο νόμος που απαγορεύει την διπλή φορολογία. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα για τους υπόχρεους μιας φορολογικής ρύθμισης επί Πολλά θέματα εσωτερικά της Γαλλίας, ε, οπότε στην ΣΕΠΕΡ, δηλαδή την Γαλλική Αρχή ε, που εποπτεύει τα φορολογικά, να συνοηθεί με τις τράπεζες όσον αφορά τις ε, συμβάσεις που συνάπτουν μεταξύ τραπεζών και των εμπλεκομένων προσώπων. Στόχος μας είναι να σταματήσει η δυσμενής διάκριση ε, σε σχέση με τις τράπεζες στην χώρα μας. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρξει κάποια ε, λύση αμοιβαία σε σχέση με τον Αμερικάνικο νόμο. Φάτκα. Βέβαια είναι και θέμα ε, σε συσχετισμού δυνάμεων. Δυνάμεων τόσο να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος στο μέλλον. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιάννησεν. Και εσείς έχετε 10 λεπτά. Καλώς ορίσατε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους ε, του Υπουργού Νέλ που δεν μπορεί να είναι παρόν εδώ σήμερα. Ε, επικροτεί όμως πολύ την διαξαγωγή αυτής της ακρόασης, διότι χρειάζεται δράση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο θέμα αυτό υπήρξε ιδιαίτερα ενεργός πάνω στο θέμα αυτό και καταλαβαίνουμε την αγανάκτηση της ομάδας αυτής. Ε, κατέλαβε λοιπόν προσπάθειες ε, απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείες και τις τράπεζες ε, των κάτω χωρών όσον αφορά αυτούς τους καταλάθους Αμερικανούς, accidental Americans. Πού βρισκόμαστε λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή. Ε, ένα ε, παγκόσμιο πρόβλημα είναι το αποκλίνον σύστημα το φορολογικό των Ηνωμένων Πολιτειών που βασίζεται στην υπηκότητα. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει κανείς Αμερικανός πολίτης ε, με τη γέννησή του, ε, σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι ε, απαιτείται να καταβάλουν φόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πολύ χαλαρούς συνδέσμους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νομοθεσία ΦΑΤΚΑ δημιουργεί προβλήματα και στη δική μου χώρα και θα ήθελα ε, να πω ότι δεν είναι μόνο το ΙΚΑ που δημιουργεί προβλήματα. Ε, υπάρχει το θέμα της ε, διαβίβασης πληροφοριών από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την νομοθεσία ΦΑΤΚΑ, οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλουν πληροφορίες για όσους ε, κατέχουν ε, λογαριασμό και συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός είναι. Εάν δεν υποβάλλεται Εάν δεν υποβάλλεται ο αριθμός TIN, ε, υποβάλλεται τα στοιχεία στο IRS χωρίς ε, τον αριθμό TIN. Ε, λογαριασμοί ε, με χαμηλά ποσά δεν χρειάζεται να ε, αναφέρονται, αλλά αυτή τη στιγμή απειλούνται οι κάτοχοι λογαριασμών ε, ότι θα απορριθούν από τις τράπεζες εάν δεν υποβληθεί ο αριθμός ΕΤΗΝ, διότι φοβούνται ότι θα επιβληθούν τεράστιες κυρώσεις, ε, κάτι που θα καταστήσει τις τράπεζες αυτές αδύνατες, θα καταστήσει αδύνατον για τις τράπεζες αυτές να δραστηριοποιούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε λοιπόν ε, πολίτες ε, στις κάτω χώρες που δεν είχαν ποτέ διαβατήριο αμερικανικό, ε, δεν έχουν την και γενικά δεν έχουν σχεδόν καθόλου σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διστάζουν λοιπόν να ζητήσουν την και να το υποβάλουν στις τράπεζές τους. Επιπλέον φαίνεται να είναι και πολύ δύσκολη η διαδικασία απόκτησης αριθμού την. Και επίσης ε, η υποβολή φορολογικής δήλωσης στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι μια διαδικασία ε, πολύ επαχθής. Ε, πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια συμβούλων οι άνθρωποι που πρέπει να το κάνουν αυτό και είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία που θα οδηγήσει και στην καταβολή φόρων στις ΗΠΑ. Έχουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα Ε, για κάτι που ε, στο 90% των περιπτώσεων ε, θα είχε μηδενικό αποτέλεσμα. Οι τράπεζές μας στις κάτω μας έχουν πει ότι έχουν 4.000 ανθρώπους με διπλή υπηκότητα χωρίς σετίν αλλά ελάχιστοι από αυτού έχουν λογαριασμό με παραπάνω από 50.000 δολάρια. Οι τράπεζες απειλούν κάποιου από αυτού τους κατόχους λογαριασμών ότι θα απορριφθούν από την τράπεζα εάν δεν υποβάλουν την. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι λόγω της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τράπεζες υποχρεούνται να προσφέρουν τη δυνατότητα λογαριασμού σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κάτω χώρες ε, λοιπόν ε, τι έχουν κάνει. Όπως ε, σας είπα, ο Υπουργός μας ήταν ιδιαίτερα δραστήριο στο θέμα αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Ξεκινήσαμε ήδη το 2006 με δύο επιστολέ, το 2016 με επιστολές προς το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κάτω χώρε μαζί με την Γαλλία νομίζω ότι είναι οι κύριοι είναι οι χώρε που κατέχουν ηγετική θέση στην κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Όπως υπόθηκε, συντάσσεται αυτή τη στιγμή νέα κοινή επιστολή από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ελπίζουμε να σταλεί σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υπουργό μου έχει σε επαφή επανειλημμένα με την ε, Ολλανδική Ένωση Τραπεζών και του έχει καλέσει προ το παρόν να μην κλείσουν λογαριασμούς ε, των ε, ανθρώπων αυτών με διπλή υπηκότητα. Επιπλέον, ε, ο Υπουργό μας επισκέφθηκε τον Μάιο ε, τη τι Ηνωμένε Πολιτείε και το βασικό αντικείμενο τη επίσκεψή του ήταν η νομοθεσία ΦΑΤΚΑ. Ήμουνα και εγώ παρόν. Συνομίλησε λοιπόν με το IRS, με τις φορολογικές αρχές και κατέστησε σαφές ε, ότι αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα οι άνθρωποι με διπλή υπηκότητα ε, στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η υποβολή φορολογικής δήλωσης στις Ηνωμένε Ε, Κάλεσε λοιπόν τις Ηνωμένε Πολιτείε να κάνουν πιο απλή, λιγότερο δαπανηρή τη διαδικασία ή να επιτρέψει στους ανθρώπους αυτούς να επεμπολίσουν την αμερικανική υπηκότητά τους με πιο εύκολο τρόπο. Ταυτόχρονα και αυτός και η δική μου ομάδα, οι δικοί μου συνεργάτες είχαμε επαφές με το IRS και με την ε, πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε συνεχείς επαφές. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Πρώτα λοιπόν έχουμε πετύχει να έχουμε μια μεταβατική περίοδο ε, για το 2017, 18 και 2019. λίγη δηλαδή αυτή η μεταβατική περίοδος. Ε, κατά την περίοδο αυτή δεν ήταν απαραίτητο να υποβάλει το αριθμός την. Έχουμε τώρα ερωταπαντήσεις από το IRS που δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν ε, προβλέπεται να επιβληθούν κυρώσεις. Αυτό θα γίνει από το 2023. Και σε περιπτώσεις ανησυχιών ε, των Ηνωμένων Πολιτών επειδή δεν υπάρχει αριθμός σε τίνη, οι τράπεζες θα έχουν ε, επαρκές χρονικό διάστημα για να επαναρθώσουν την κατάσταση. Πιστεύουμε ότι αν οι τράπεζε κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκτήσουν ε, του τους αριθμούς ετήν που τους ε, λείπουν, ε, θα είναι δυνατόν. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ νωρί να κλείσουν αυτή τη στιγμή τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι φορολογικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών είπαν ότι εάν απεμπολίσει κανείς την αμερικανική υπηκότητα θα απαλλαγούν και από τις υποχρεώσεις αυτές ε, και αυτό θα ισχύσει και ε, για ε, άλλους υπηκόους των ΗΠΑ με διπλή υπηκότητα. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Προξενείο στις κάτω χώρες, Έχουμε θεσπίσει το σύστημα εάν κάποιος ε, ξεκινήσει τη διαδικασία ε, αυτήν ε, λαμβάνει σχετικό πιστοποιητικό το οποίο μπορεί να δείξει στην τράπεζά του οπότε η τράπεζα καταλαβαίνει ότι δεν απαιτείται αριθμό ΕΤΗΝ. Πιστεύουμε ότι τα αποτέλεσματα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα ήταν χρήσιμα, αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα βοηθήσουν τι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, τι ε, Τράπεζε ε, και τους Ιδιώτε, Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επιθυμητικό αποτέλεσμα. Το, το επιθυμητό αποτέλεσμα θα ήταν η τροποποίηση του φορολογικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο όμω δεν βλέπω να συμβαίνει βραχυπρόθεσμα. Η συμβουλή μας λοιπόν προς ανθρώπους με διπλή υπηκότητα είναι να ενεργήσουν γρήγορα ώστε να επιλέξουν είτε να πεμπολίσουν την ε, αμερικανική τους ε, υπηκότητα για να απαλλαγούν από όλες αυτές τις διαδικασίες ή εάν επιθυμούν να παραμείνουν υπήκοοι των ΗΠΑ ε, να αποκτήσουν αριθμό την. Έχουμε ακόμη κάποια θέματα που μας απασχολούν, τα οποία θα ε, αναφέρουμε απέναντι στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, ένα από αυτά είναι ότι τα τέλη απεμπόληση τη ε, υπηκότητα είναι 2.000 ευρώ, ε, παλιότερα ήταν 450 δολάρια, θα πρέπει να χαμηλώσει λοιπόν ε, το τέλο αυτό. Δεύτερον, για να υποβάλει κανεί φορολογική δήλωση, δεν θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο το σύστημα αυτό. Προτείνουμε λοιπόν απαλλαγή στις ε, περισσότερες ε, περιπτώσεις να απλοποιηθεί το σύστημα και το άλλο που ζητάμε από τις ΗΠΑ είναι να φροντίσει οι τράπεζες να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να μην επιβληθούν σε αυτές κυρώσεις, διότι αυτό ε, θα τις κάνει πιο ανοιχτές απέναντι στους ανθρώπους με διπλή υπηκότητα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να επισημαίνουμε τα θέματα που μας απασχολούν, ε, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για όσα τόσο ξεκάθαρα μας τα είπατε και τώρα ο κ. Κάζερ έχει το λόγο και αυτός για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ αρχικό στο ζήτημα της φορολογικής συμμόρφωσης. Την τελευταία δεκαετία η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης έχει καταστεί βασική προτεραιότητα για κυβερνήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής και φορολογικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί σήμερα σημαντικότατο το θέμα στην μέσα διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίση. Η ΦΑΤΚΑ, που είναι ο νόμος περί φορολογικής συμμόρφωσης των Ηνωμένων Πολιτειών και οι μετέπειτα διακυβερνητικές ε, συμφωνίες έχουν ως στόχο να καταπολεμήσουν την ε, φοροδιαφυγή από αμερικανική σκοπιά. Η ΦΑΤΚΑ στοχεύει σε Αμερικανούς φορολογουμένους πολίτες οι οποίοι κρύβουν περιουσιακά στοιχεία σε offshore εταιρείε ε, και προσπαθούν να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους στη χώρα τους. Η ΦΑΤΚΑ βασίζεται σε ενδιάμεσους συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστικών ιδρυμάτων και άλλων ξένων φορέων. Με δύο λόγια, η ΦΑΤΚΑ επιβάλλει δύο βασικές κατηγορίες απατήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πρώτον, ένα χρηματοπιστικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να εξετάζει την πελετική του βάση με βάση όλες τις δέουσες διαδικασίες προκειμένου να προσδιορίσει τυχόν ανακοινωτέους ε, λογαριασμούς στις ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων πολιτών των ΕΠΑ αλλά και νομικών προσώπων που ελέγχονται με βάση την, ε, την ε, αμερικανική νομοθεσία. Επίσης, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει τα ευρήματά του στις ε, αμερικανικές αρχές μέσω των εγχώριων φορολογικών αρχών. Πέρα από αυτά, η ΦΑΤΚΑ αποτέλεσε καταλήτη για την ανάπτυξη της ε, διεθνούς ε, ανταλλαγής πληροφοριών και του αντίστοιχου συστήματος που αναπτύχθηκε στη βάση του CRS του ΟΣΑ και της αναθεωρημένης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διοικητική συνεργασία. Συνολικά, η ΦΑΤΚΑ, οι διακυβερνητικές συνεργασίες και όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα συναποτελούν ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί ένα διεθνές σύστημα φορολογικής αναφοράς το οποίο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής. Ως ε, Ομοσπονδία Τραπεζών της Ευρώπης, εμεί υποστηρίζουμε την καταπολέμηση της φορολογική απάτης. Οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τον νόμο και να τηρούν τους κανόνες σχετικά με τη φορολογία. Συγκεκριμένα, μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ ή που εμπορεύεται αμερικανικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κίνδυνο ε, να θεωρηθεί μη ε, συμμορφούμενο γιατί ε, μπορεί να, ε, επιβληθεί, να του επιβληθεί ποινή 30% παρακράτησης ε, φόρου για όλα τα εισερχόμενα εισοδήματα. Τα τελευταία 10 χρόνια η Ομοσπονδία μας επιδίδεται σε έναν επικοδομητικό διάλογο με κυβερνήσεις και με χρηματοπιστικά ιδρύματα και φορολογικέ αρχές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Διαρκώ, εφιστούμε την προσοχή του IRS και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστικά ιδρύματα και οι πελάτες τους. Προσπαθούμε πάντοτε να προτείνουμε ρεαλιστικές προτάσεις για να υπερβούμε τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες με τις εν μέρη ακόμη και αντιφατικές ε, οδηγίες που πρέπει να εφαρμόζουν από τις διάφορες ευρωπαϊκές και αμερικανικές δικαιοδοσίες. Υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τους προϋπάρχοντες ε, λογαριασμούς. Η ΦΑΤΚΑ ε, υποχρεώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξετάζουν την πελιατική τους βάση ώστε να προσδιορίζουν σε ε, εύθετο χρόνο ε, λογαριασμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανακοινωτέοι προς τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ. Αν στη βάση κριτηρίων που έχουν ε, προσδιορίσει οι ίδιες οι ΗΠΑ. Όταν βρίσκεται ένας τέτοιος λογαριασμός θα πρέπει αυτόματα να διαβιβάζονται οι σχετικέ πληροφορίες στι Αμερικανικέ Φορολογικέ Αρχέ, εκτό αν έχει λάβει από τον ε, κάτοχο του λογαριασμού ρητή δήλωση ότι δεν είναι Αμερικανό πολίτη. Σε περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν αναφέρει στις φορολογικές αρχές ένα τέτοιο λογαριασμό, τότε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί μη συμμορφούμενο και να του επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις. Λόγω αυτής της κατάστασης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά από δύσκολες καταστάσεις. Για παράδειγμα, κάποιοι πελάτες δεν έχουν απαντήσει ποτέ στα ερωτήματα που τους απευθύνει η τράπεζά τους ή έχουν απαντήσει ότι είχαν δυσκολία να αποκτήσουν αριθμό φορολογικού μητρώου στη ΣΥΠΑ. Και αυτό αφορά κυρίως τους κατατύχει Αμερικανούς, εκείνοι οι οποίοι έλαβαν την Αμερικανική υπηκότητα με βάση το δίκαιο των ΗΠΑ, γιατί γεννήθηκαν στις ΗΠΑ και έφυγαν σχεδόν αμέσως, οπότε έχουν ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους εκτός ΗΠΑ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις πολύ βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες γιατί τους ζητείτε να έχουν αφημί αμερικανικό. Άλλο πρόβλημα είναι ότι κατά το άνοιγμα λογαριασμού ο πελάτης πρέπει να υπογράψει μια αυτοπιστοποίηση και αν τόπος γέννησης είναι περιοχή των ΗΠΑ, πρέπει να επιβεβαιώνει αν είναι ή όχι αμερικανικός ε, πολιτής. Σε περίπτωση που είναι θα πρέπει να δίνει αμερικανικό αφημί ή διαφορετικά μπορεί να δηλώνει ότι δεν είναι αμερικανός πολίτης, περίπτωση κατά την οποία θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού απώλειας της αμερικανικής Ιθαγένειας που έχει λάβει ή εύλογη αιτιολόγηση για το γιατί δεν διαθέτει τέτοιο έγγραφο στα χέρια του. Να προσπαθήσω τώρα να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Σχετικά με τις τελευταίες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, και επιτρέψτε μου να σας δώσω και κάποιες συστάσεις από την πλευρά μας. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών έπειτα από συστάσεις της οδήγησε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει το σημείωμα 2017-46, το οποίο παρέχει μια περίοδο χάριτος που εκπνέει τον επόμενο μήνα και που είχε διάρκεια τρία έτη. Στη διάρκεια αυτών των τριών ετών, η μη υποβολή αφημί Αμερικανικού δεν επιφέρει αυτόματα απώλεια του καθεστώτος του συμμερφούμενου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες προϋποθέσεις. Το ξένο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να δώσει ημερομηνία γέννησης του πελάτη και ετησίως να ζητεί ε, αμερικανικό αφημί. Όπως είπα, η περίοδος χάριτος αυτή εκπνέει σύντομα. Και γι' αυτό το λόγο επισκεφτήκαμε την Ουάσιγκτον αρκετές φορές φέτος, εντός του 2019, και αποστήλαμε και μια σειρά από επιστολές. Και στα μέσα Οκτωβρίου, με χαρά θα πω, διαβάσαμε ένα σημείωμα από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, με την μορφή συχνών ερωτήσεων όπου καταφέραμε να διαβάσουμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας ανακούφισαν και μας καθυσίχασαν σε έναν βαθμό. Δυστυχώς όμως το έγγραφο αυτό δεν έχει κάποιον επίσημο χαρακτήρα, δεν είναι επίσημο έγγραφο, περιέχει ασάφειες και το Τραπεζικό Ίδρυμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια σαφή επίσημη παρα, παράταση αυτής της περίοδου χάριτος. Ιδανικά βεβαίως θα θέλαμε και μια μόνιμη λύση. Επίσης, χρειαζόμαστε παράταση για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται υπό το μοντέλο IGA2. Χρειαζόμαστε λύση για τους νέους λογαριασμούς και τις συναφείς διαδικασίες. Ελπίζουμε λοιπόν οι Αμερικανικές αρχές να επιδείξουν ε, προθυμία να ξανανοίξει συζήτηση σχετικά με τις ε, IGA τις διακυβερνητικές αυτές συμφωνίες. Αυτά από μένα και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για τα όσα μας είπατε και τώρα έχουμε τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις από πλευρά των βουλευτών. Ποιος θέλει το λόγο? Η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους αναφέροντες και τους ε, κατατύχει Αμερικανούς, τους Accidental Americans ε, που ε, ήρθαν εδώ στο Κοινοβούλιο σήμερα το πρωί. Καταλαβαίνω πολύ καλά την αγανάκτηση των ανθρώπων αυτών. Συζητάμε τα θέματα αυτά εδώ και χρόνια, θέτοντας συνεχώς τα ίδια ερωτήματα. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτήν την προθεσμία, όπως ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών. Η δράση κάποιων κρατών μελών ε, πρέπει να επενεθεί, αλλά η αδράνεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι απογοητευτική. Νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και να είμαστε απόλυτα σαφείς. Καταλαβαίνω πολύ καλά τις υποθέσεις αυτές. Εγώ είμαι κατά τύχη Τανζανιανή και αναρωτιέμαι ποια θα ήταν η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν μιλούσαμε για πολίτες άλλης χώρας από της ευρωπαϊκή Ένωσης, εάν θα υπήρχε άλλη νοοτροπία, άλλη στάση στα θέματα αυτά. Αυτό είναι μια επιπλέον δυσκολία για πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς. Σε λίγους μήνες λοιπόν, σε λίγες εβδομάδες, σε λίγη αυτή η προθεσμία και ακούσαμε ότι γίνονται συζητήσεις εντός του Συμβουλίου για ανάληψη κάποιας βασικής δράσης. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής ε, Νομοσπονδίας Τραπεζών, διότι ε, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει σαφής παράταση. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο άνοιγμα, διότι όπως υπόθηκε στην αρχή, όπως είπε στην αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει εδώ και χρόνια, ασκεί εδώ και χρόνια πίεση Τι πιστεύετε ότι απαιτείται ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, να ενεργήσουν ε, ε, πολύ πιο στεναρά. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς τους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ, ο Πίτερ Γιάρ. Ευχαριστώ. Και εγώ. Τους αναφέροντες και τους εμπειρογνώμονες που βρίσκονται εδώ στην ακρόασή μας σήμερα. θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα την ε, κατάσταση και έχω κρατήσει εδώ σημειώσεις, ε, έχουμε το γενικότερο πλαίσιο, έχουμε την ε, καταπολέμηση της απάτης, χρειάζεται ροή των πληροφοριών, πολύ σωστά όλα αυτά. αλλά υπάρχει ένα ρητό ότι στο ρεύμα ε, της αλήθειας ε, κολυμπάει και το ψέμα. Ε, πολύ ωραία λοιπόν όλα αυτά που κάνουμε, αλλά υπάρχουν και παράπλευρες ε, απώλειες ή δυσκολίες, ε, τις οποίες δεν υποψιάζεται κανείς στην αρχή. θα πρέπει να δεχτούμε ότι η κάθε χώρα αναπτύσσει το δικό της φορολογικό δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει αυτό και ε, το, οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν το ίδιο. Το τρίτο θέμα που με απασχολεί ωστόσο είναι το εξής. Ε, είναι γνωστό το θέμα γιατί δεν έχει λυθεί βλέπουμε ανθρώπους που έχουν γίνει θύματα της ε, σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για φορολογικό δίκαιο, η Κομισιόν λέει συγγνώμη, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μια απόφαση με ομοφωνία, αλλά εδώ πέρα είναι χίλια δυο άλλα θέματα μέσα. Έχουμε την προστασία των δεδομένων, έχουμε το θέμα της ηθαγένειας, έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είναι λοιπόν αρμόδια για τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε θέμα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μήπως ε, θα έπρεπε ε, οι ε, πρωθυπουργοί, οι Κομισιόν να παρουσιάσουν το θέμα απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Η ερώτησή μου πάντως είναι η εξής. Είναι πράγματι απίστευτη η κατάσταση αυτή. Είναι ανήκουστο το θέμα, πράγματι, συμφωνούμε σε αυτό. Η ερώτησή μου είναι ποια θα ήταν τα βασικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Εγώ έχω καταγράψει εδώ πέρα δύο, αλλά πείτε μας ποια είναι τα βασικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Εάν ε, δεν έχω καταλάβει σωστά, παρακαλώ να μου το πείτε, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι απαραίτητο είναι καταρχάς να έχουμε μία συμφωνία κυρίων κατά τη μεταβατική περίοδο και να παραταθεί αυτή τώρα που λύγει. Και επίσης, ε, εάν κάποιος επιθυμεί να παραιτηθεί από την ε, αμερικανική του υπηκότητα, να μπορεί αυτό να γίνει με τρόπο απλό και πιο οικονομικό. Υπάρχουν ε, άλλα μέτρα που πιστεύετε ότι θα πρέπει να ληφθούν. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Η κυρία Ίντβελτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές μας σήμερα. Εγώ δεν έχω να σας απευθύνω κάποιο ερώτημα συγκεκριμένο τα, τα, ερωτήματα που όλοι μας ε, έχουμε είναι ερωτήματα που απευθύνονται στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν. Και εδώ κάνω βεβαίως εξαίρεση ρητή για τη Γαλλία και τις ε, κάτω χάρες που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών τους. Όμως τα άλλα 26 κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απουσιάζουν, υπόπτως μάλιστα. Και κάθε φορά που διαβάζω την απάντηση ε, τις απαντήσεις μάλλον του κυρίου Μοσκοβισή ε, είναι πραγματικά προσβλητική οι προσβλητικές οι απαντήσεις του γιατί ε, έχει κανείς την, την αίσθηση ότι τον ενδιαφέρει να προστατεύσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις φορολογικές αρχές των ΙΠΑ και όχι τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι, έχουμε δικαιώματα τα οποία πρέπει και να τα υπερασπιστούμε αυτό που γνωρίζω είναι το ζήτημα αυτό είχε ε, υποπέσει στην αντίληψή μου το 2012. Γιατί, Γιατί οι γαλλικέ τράπεζε είχαν επισημάνει τότε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι του ασκείται πίεση. Και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να διαπραγματευτεί μια διευθέτηση του ζητήματο με του Αμερικανού, όχι για να προστατεύσει πάλι τους, ε, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά για να προστατεύσει τι τράπεζε. Καλώ, αλλά. Ε, τι να πω, ακόμη και αυτό το έχουν εγκαταλείψει πια. Ελπίζω αυτή η γεωπολιτική μεταστροφή που έχει ανακοινώσει η Ursula von der να μας οδηγήσει επιτέλους σε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί από τις εθνικές πολιτικές οι εθνικές αρχές δεν φαίνεται να γίνεται και τίποτα. Υπάρχουν κάποιες ε, προτάσεις για βραχυπρόθεσμη ανακούφιση του και ε, επίλυση του ζητήματος. Εγώ διαπιστώνω όμως ότι και πάλι το βάρος το επομίζονται τα άτομα που επηρεάζονται άμεσα, είναι πραγματικά εξαιρετικά ενοχλητικό το γεγονός ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις και οι Κομισιόν προκρίνουν τις διατλαντικές σχέσεις έναντι των, των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Αποδέχονται και μάλιστα το κάνουν σε πολλούς τομείς πολιτικής ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ισχύει και εφαρμόζεται εδώ. Ε, κύριε Γιάρ, ναι, ορθώς είπατε ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα να θεσπίζει την νομοθεσία της συμπεριλαμβανομένη φορολογική. Ταυτόχρονα όμω η ΕΠΑ και η Ερυθρέα είναι οι, δύο, οι μόνε δύο χώρε που έχουν φορολογικό σύστημα βάση ηθαγένεια. Εμεί είμαστε υπερδύναμοι οικονομικοί. Μπορεί κάποιο να μου εξηγήσει γιατί δεν χρησιμοποιούμε την ε, ε, δύναμη 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καταναλωτών για να πείσουμε τους ε, ε, Αμερικανούς, τουλάχιστον να κάτσουν στο τραπέζι, των, στο τραπέζι διαπραγματεύσεων μαζί μας. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο το ζήτημα της ΦΑΤΚΑ και, τον, και τους κατατύχει Αμερικανούς. Πρόκειται θεμελιωδώς για τις διατλαγικές σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είμαστε αδύναμοι αυτή τη στιγμή, διότι 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Όχι απλά πρακτικό πρόβλημα, είναι ένα ουσιώδε πολιτικό πρόβλημα. Οπότε πρέπει να ασκήσουμε όσο μεγαλύτερη πίεση γίνεται. Μετά από 8 χρόνια φάτκα, καταλαβαίνω πλήρω την ε, δυσαρέσκειά σα και τη δυσφορία σα για την έλλειψη ε, προόδου το ότι δεν έχει σημειωθεί κανένα, καμία πρόοδος, ε, με εξαίρεση τις γαλλικές και ολλανδικές αρχές, αλλά πραγματικά νομίζω ότι πρέπει και ως Επιτροπή να ε, πάμε στην Φιλανδική Προεδρία ώστε να την πιέσουμε επιτέλους να μιλήσει με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους Αμερικανούς. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αν συμφωνείτε, τώρα να δώσουμε δύο λεπτά σε κάθε έναν ε, από τους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν στα όσα είπαν και ερώτησαν οι βουλευτές. Έχετε το λόγο. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, ο κύριο Μαρέ, ο κύριος Μαρτέν, συγγνώμη, ο κύριο Γιάννη, ο κύριο Κάιζερ. Δεν πειράζει. Καλά, με την ίδια σειρά. Γιάννη, εσεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι απευθύνθηκε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση προς εμένα, αλλά θα ήθελα εγώ από την πλευρά μου να κλείσω λέγοντας ότι καταλαβαίνω πολύ καλά την αγανάκτηση ε, με το ε, φορολογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει βράχη πρόθεσμα. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε γρήγορες λύσεις. Πετύχαμε κάποιες από αυτές. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, έχει γίνει σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι σημαντικό σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη και με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουμε τις ενέργειές μας απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείες Θα πρέπει να μειωθεί δηλαδή το τέλος ε, για ε, την απαλλαγή από την ε, αμερικανική υπηκότητα και σε πολλές περιπτώσεις να, να υπάρχει απαλλαγή υποχρέωσης της υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάζερ, εσείς που είχατε και πιο πολλές ερωτήσεις που σας απευθύναν. Αν κατάλαβα καλά εγώ τις ερωτήσεις, Ε, πόσο εύκολο είναι να πετύχουμε παράταση από τι ΗΠΑ. Ε, δεν είναι πολύ εύκολο να το απαντήσω αυτό, διότι πίσω από όλη αυτή την ε, συζήτηση έχουμε τον φορολογικό κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αποκλίνουν από αυτόν. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές τράπεζες, η βασική μου ανησυχία είναι το θέμα της συμμόρφωσης Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Υπάρχουν κάποιες θετικές πλευρές. Υπάρχουν κάποια θετικά μηνύματα. Όπως γνωρίζετε έχει υποβληθεί νομοσχέδιο στο Κογκρέσο Κάποιοι πολιτικοί λοιπόν στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, ανησυχούν σχετικά με την κατάσταση. Οι ερωταπαντήσεις ε, που δημοσιεύτηκαν ε, στις 15 Οκτωβρίου ήταν πολύ θετικό σημάδι και εμείς ως Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Όσον αφορά τις γρήγορες λύσεις, χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια δικαίου. Οι τράπεζες ανησυχούν ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικό κίνδυνο να θεωρηθούν να θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται. Αυτό λοιπόν ε, θα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη βεβαιότητα, ασφάλεια και θέλουμε το περιεχόμενο των ερωταπαντήσεων ε, να ε, μετατραπεί σε επίσημο έγγραφο και γι' αυτό εμείς ως Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών στείλαμε επιστολή την προηγούμενη Παρασκευή στον κύριο Νόσιμ ε, των Αμερικανικών Αρχών. μακροπρόθεσμα. Μάλλον πρέπει να ξανανοίξουμε την ε, συζήτηση ε, για τις διακυβερνητικές ε, συμφωνίες. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα με τη ΦΑΤΚΑ είναι ότι δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων του ΟΣΑ, που σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ πιο ευέλικτα. Μακροπρόθεσμα, λοιπόν, λοιπόν επιθυμούμε ξανά άνοιγμα της συζήτησης και ε, σύγκληση ανάμεσα στον ΦΑΤΚΑ και τις απαιτήσει υποβολής εκθέσεων του ΩΣΑ. Κύριο μαρτέ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα κάποια ερώτηση. Ε, Προ το πρόσωπό μου. Όμως θέλω να σταθώ στα εξή δύο. Πρώτα πρώτα να σα πενδυμίσω τη σημερινή κατάσταση. Δύο-δύο-δύο ε, θέλω να σα πω γιατί όλα αυτά έχουν συγκλονίσει το Γαλλικό Κοινοβούλιο γιατί έρχονται σε ε, αντίθεση με την κουλτούρα μας, το πνεύμα που μας διαπνέει. Αυτές οι εγγύσεις, δηλαδή είπαμε ότι Υπάρχει η οδηγία πάντου του 14 που δίνει δηλαδή κάποιες ε, εγγύησεις σε όλους όσοι νομιώς διαμένουν στην ε, Ένωση να έχουν κάποια δικαιώματα όσον αφορά τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και να ανοίξουν ένα λογαριασμό στη Γαλλία. Οπότε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι τερατώδες και επίσης το ότι σήμερα ε, έχουμε τις τράπεζες να ε, δίνουν τα δεδομένα αυτών των προσώπων χωρίς την ένεσή τους στους Αμερικανούς. Ε, αυτό έρχεται σε σύγκρουση με ε, τον σχετικό κανονισμό για τα δεδομένα. Οπότε έχουμε όλες αυτές τις ε, νομικές παρανοήσεις, τους παραλογισμούς. Θα πρέπει αυτά πρώτα-πρώτα να αρθούν. Και κάτι άλλο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το θέμα της αμοιβαιότητας. Ήμασταν η πρώτη χώρα το 2014 που ψηφίσαμε την διακυβερνητική συμφωνία κυρώθηκε στο Κοινοβούλιο στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και διάβασα τα πρακτικά της συνεδρίας εκείνης και ο κ. Γκαλή που ήταν ο εισηγητής και ε, διαμακρόν εξήγησε στους Γάλλους ότι μόνο επί της βάση ισχύει αυτή η συμφωνία ότι δηλαδή θα ισχύει το ίδιο και για τους ε, ε, ε, Γάλλους εκπατρισμένους στην Αμερική σε σχέση με τη γαλλική φορολογία. Οπότε βέβαια ε, πρέπει να έχει γίνει και κύρωση από τους Αμερικανούς. Δηλαδή ήταν μια υπόσχεση που έπεσε στο κενό. Άρα δεν ήρθε αυτό το νομικό κενό ότι δηλαδή ότι θα πρέπει να εξισορροπήσουμε, να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των ΗΠΑ ε, και της Ευρώπης. Άρα αυτό είναι πολύ απογοητευτικό το πώς γίνονται τα πράγματα και πώς υφιστάμεθα όλες αυτές τις αρνητικές συνέπειες ενώ μιλούμε για το Αμερικανικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ότι ήμασταν οι μόνοι εμείς που προσυπογράψαμε αυτές τις διακυβερνητικές συμφωνίες είπα και κρατών μελών οπότε ό, κάποια στιγμή θα πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι να ξυπνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε όλα τα μέλη του πάνελ, όλους σας. Ε, ευχαριστώ για όλα αυτά τα δημιουργικά, τα θετικά μας είπατε. Α, ο Θέλω να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα και ένα αίτημα προς την Ένωση Τραπεζών. Είπαν εισηγητικά ότι η ΦΑΤΚΑ εντάσσεται στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όμως, η ΦΑΤΚΑ εξυπηρετεί μόνο τα αμερικανικά συμφέροντα, όχι τα ευρωπαϊκά. Δεν θα ήταν λογικό οι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε να πούν ποιο είναι το κόστος που επομίζονται οι ευρωπαϊκές Τράπεζε για την υπεράσπιση των ε, αμερικανικών φορολογικών συμφερόντων. Αν τα συνδυάσετε όλα τα κόστη που καταβάλουν οι ευρωπαϊκές Τράπεζε είναι δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ε, γιατί δεν αξιοποιούμε όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί μάλιστα από το 2012, και να το χρησιμοποιήσουμε ως επιχείρημα ότι είναι ένα τεράστιο ποσό το οποίο ε, καταβάλουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες στην ουσία για την υπεράσπιση των αμερικανικών φορολογικών συμφερόντων. Νομίζω ότι θα ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό επιχείρημα αυτό. Le doy la palabra para que conteste a esta pregunta. Daríamos por cerrado este Ωραία, το έκλεισε μέσα αυτό το πάνελ και έχουμε τώρα το, τη δεύτερη ομάδα εργασίας, το δεύτερο πάνελ, αλλά προσοχή 12.30 δεν θα έχουμε διερμηνία. Παρακαλώ ένα λεπτό για την απάντηση αυτή τη ερώτηση τα το μέλη του πρώτου πάνελ. Πολύ σύντομα θα απαντήσω. Φυσικά, το κόστος συμμόρφωσης αποτελεί βασικότατο επιχείρημα που έχουμε χρησιμοποιήσει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεών μας. Από την αρχή μάλιστα. Yeah, but the system is in place now. No entremos en debate. Μην ανοίξουμε συζήτηση όμω. Καλώ λέει πρόεδρο. Οπότε, κλείνει αυτό το πάνελ. Ευχαριστώ τον αναφέροντα. Αναφέρουμε και του ε, εισηγητέ και του βουλευτέ για τα όσα ενδιαφέροντα είπαν. Πάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Εδώ έχουμε τον Φαμπιέν Λεάγκερ που είναι πρόεδρος του φορέα της Ένωσης, του Σωματείου τέλος πάντων αυτών των ε, συμπτωματικά Αμερικανών. Επίσης τον Φίλιππο Νοσέδα που είναι καθηγητής στο King's College του Λονδίνου, την Ελίσσα Φέικεμαν από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ισμήρη Ριγοπούλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασία Δεδομένων. Λεάγκρε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, Μισό λεπτό, μισό λεπτό, λέει η πρόεδρο, διακόπτη. Αντί για 10, Σα κόβω στα 8, για να υπάρχει χρόνο να έχουμε διερμηνία για όλου. Συνέχεια. Σας ε, θέλω να σας πω για του ε, Αμερικανού, του οποίους εκπροσωπώ ότι πρώτα πρώτα σα ευχαριστούν για την ευκαιρία αυτή που μα δώσατε να σα πούμε με λεπτομέρειε το τι έχει γίνει από την κοινωνία των πολιτών. Σε ευχαριστώ την Τζουντ που ξεκίνησε αυτή την αναφορά, ε, τον Τζουντ συγγνώμη, ε, εκείνη μάλλον, συγγνώμη, συγγνώμη, ε, και γι' αυτό ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και η απόκριση του Ευρωπαϊκού και δεν είναι δυνατόν να είμαστε αποτελεσματικοί χωρίς να έχουμε κάποιον φορέα και γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το σωματείο των κατατύχει Αμερικανών τον Μάη του 2017 και θα επανέλθω σε αυτό που έχουμε κάνει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενεργήσουμε τι θα πει ένας τυχαίος, ένας ομιλικός Αμερικανός είναι αυτοί οι οποίοι τυχαία ε, λόγω της γέννησής τους ε, κληρονόμησαν την ηθαγένεια αλλά δεν έχουν κάποια επαφή με τις ΗΠΑ, δεν έχουν μείνει, δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν σπουδάσει περισσότεροι, δεν έχουν καν ε, ε αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε χρησιμοποιώντα τα νομικά ότι είναι κάποιοι πολίτες που δεν πληρούν κάποια κριτήρια του ε, αμερικανικού νόμου, του αμερικανικού δικαίου, τόσο ώστε κάποιος να μπορεί να ε, διαβιβάσει την ε, ηθαγένεια. Και γι' αυτό πρόκειται για κάποιους οι οποίοι έχουν ζήσει τουλάχιστον πέντε χρόνια, λέει ο νόμος, της είπα, και δύο χρόνια μετά την ηλικία των 14 και έχουμε σε αυτή την αρχή ε, τη φορολογία επί τη βάση τη ηθαγένεια. Δηλαδή, φορολογούνται οι Αμερικανοί όποια βρίσκονται στον κόσμο, οπότε θα πρέπει κάθε τέτοιος συνολικό Αμερικανό να δηλώνει τα εισοδήματά του και τους ε, λογαριασμού του στι φορολογικέ αρχέ. Μέχρι το 2014, ε, οι τυχαία Αμερικανοί αγνοούσαν το ότι έχουν φορολογικές υποχρεώσεις γι' αυτό ε, θεωρούσαν ότι είναι απλώς ε, ένα κληροδότημα ε, η Θαγένεια χωρίς να έχει νομική σημασία. Δεν είχαν επαφή με την Αμερικανική δίκηση και δεν είπαμε δεν είχαν και καμία κάλυψη κοινωνικής πρόνοιας. Οπότε το 2014 όπως τα περισσότερα κράτη-μέλη η Γαλλία ε, προσυπέγραψε αυτή την ε, συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, ούτω ώστε παντού να ισχύσει και για τις γαλλικές τράπεζες ε, ο νόμος ΦΑΤΚΑ. Και είχαμε το IGA που είναι η εφαρμογή αυτής της διεθνούς συμφωνίας που σήμαινε ότι όλα τα δεδομένα τα σχετικά πήγανε στη ΣΥΠΑ από τη Γαλλία. Και από το 2014 οι τράπεζες άρχισαν να απευθύνονται ε, και να ασχολούνται με τους πελάτες τους που είχαν στοιχεία ε, αμερικανικής ηθαγένειας. Τους ζήτησαν να συμπληρώσουν κάποια έντυπα και τους είπαν ότι θα πρέπει να έχουν ε, κάποια πιστοποιητικά, να απεμπολίσουν την ηθαγένεια και πρόκειται επομένως για κάποιους που είχαν κάποιον κωδικό, είναι αυτή η τυχαία Αμερικανή που γίνεται μετά το 1986. Το ίδιο έγινε και στα κράτη-μέλη που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία και η προεδρική ε, η Προεδρία της Μάλτας το 2017 ε, έρθε σε συνεννόηση με τις Αμερικανικές Φορολογικές Αρχές σε σχέση με αυτό τον κωδικό SSN ε, και 31 Δεκεμβρίου εξέπνευσε η μεταβατική προθεσμία και μετά την 1η ε, Πρώτου του 20 και πάλι θα πρέπει ε, να έρχονται σε συνεννόηση οι γαλλικές τράπεζες και ακόμη και αν οι φορολογικέ αρχές τώρα οι Αμερικανικές έχουν πιο πολύ ευελιξία. Είπαμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να επιβαρύνουν κατά 30% ε, τους λογαριασμούς αυτούς. Ε, και είχαμε επίσης μια ανακοίνωση στους 17 του 19 από τις γαλλικές τράπεζες που είπε ότι είναι 40.000 λογαριασμοί που θα επιβαρυνθούν και θα κλείσουν. Ε, τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα για αυτά τα πρόσωπα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να προσφύγουν κάπου κατά αυτών των τραπεζικών μέτρων. Ε, θεωρούν ότι αυτές οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ βαριές και προτιμούν να μην δεχτούν Αμερικανούς πελάτες οι τράπεζες. Και οι περισσότερες τράπεζες επομένως αυτό κάνουν. Ε, τώρα και αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχει αυτή η ηθική βλάβη εις βάρος αυτών των προσώπων και επίση είναι δυνατόν να τους επιβληθούν και κάποιες κυρώσει. Οπότε υπάρχει και χρηματική ζημία. Ε, ήδη έχουν εξοδέψει αυτά τα πρόσωπα πάρα πολλού δικηγόρου και ήδη έχουν πληρώσει κάποιου φόρου. Ακόμα και κάποιο θεωρηθεί US person, αυτομάτω, αυτοδικαίω. Ε, με το που έχει την ηθαγένεια έχει ένα σωρό συνέπειες ε, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποια τραπεζικά προϊόντα Υπάρχει δεσμενής ε, διάκριση ε, σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν αμερικανική ηθαγένεια. Οπότε αυτό που δεν θέλουμε να γίνεται είναι να σταματήσει όχι μόνο η ΦΑΤΚΑ, ε, να μην υπάρχει αυτή η εξοδευτικότητα για αυτά τα πρόσωπα. Και, και στο Βέλγιο επίσης έχει συγκροτηθεί ένας φορέας για κάποιους τέτοιους ε, τυχαίους ε, Αμερικανούς, αλλά και στη Γερμανία, στις κάτω χώρες, στην Ιταλία, οπότε υπάρχει ε, μια σημαντική εκστρατεία ενημέρωσης και τα μήμια έχουν ενδιαφερθεί, αλλά επίσης έχουμε προσβάσεις και στη δικαιοσύνη τον Οκτώβριο του 2017 κάναμε μια νομική μελέτη από τον καθηγητή Ρεζίμπι Σμιτ και προσφύγαμε στο Conseil d'État και ζητήσαμε να ακυρωθεί το σχετικό διάταγμα για την διαβίβαση των γεγονότων και είπαμε ότι δεν υπάρχει επίσης ε, αμοιβαιότητα σε σχέση με αυτή την ρύθμιση με τη ΣΥΠΑ. Και είπαμε ότι ο μηχανισμός για τα δεδομένα δεν λαμβάνει, δεν υπόψη ότι οι περισσότεροι τους οποίους θίγει δεν έχουν καμία σχέση με τη ΣΥΠΑ. Δεν προβλέπεται καμία προστασία για τα δεδομένα και έτσι δεν διορθώνονται ε, τα σφάλματα ή αστοχίες που μπορεί να συμβαίνουν το 2017. Η Μοντ ε, δημοσίευσε την περίπτωση ενός Γάλλου που γεννήθηκε στον Καναδά και στείλαν κατά λάθο τα στοιχεία του στους ε, Αμερικανούς. Επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, έκρινε στις 6 Δεκάτου του 2015 στην περίπτωση της Χρέμς ότι δεν υπάρχει επαρκής προστασία σε αυτά τα δεδομένα από πλευράς των ε, Αμερικανών. Επίσης, ε, ελπίζουμε ότι η Γαλλία τελικά θα σεβαστεί αυτή την προδικαστική ερώτηση ή θα, για τέλος πάντων θα προσφύγει, θα ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, γιατί αυτό προβλέπεται ε, με την απόφαση της τεταρτης 10 του 18. Και τελικά η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να γίνει ε, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επί παραλήψη κατά της Γαλλίας. Το Μάρτιο του 19 ο φορέας μας ε, προστάτευσε 306 τέτοιους Αμερικανούς ε, συμπτωματικούς σε σχέση με κάποια μήνυση κατά των τραπεζών για δυσμενή διάκριση. Είχαμε επίση την ε, έκθεση Λελούς Μπερζέ όσον αφορά την εξοεδαφικότητα της Αμερική νομοθεσίας και αφορούσε αυτό το πρόβλημα των τυχαίων Αμερικανών. Το Μάιο του 19 είχαμε και άλλη μια ε, έκθεση κοινοβουλευτική, την ε, έκθεση Le Fur που αφορούσε τις συνέπειες αυτής της νομοθεσίας της Αμερικανικής για την εξοδευτικότητα. Όσον αφορά τώρα αυτά τα οποία κάναμε, είπαμε ότι Θέλουμε να δούμε τι γίνεται ε, και για αυτό εγγράφηκε το θέμα στο ΕΚΟΦΗΝ. Ε, το ζήτησε η Φιλανδική Προεδρία ε, και διάφορα κράτη-μέλη είπαν ότι θέλουν να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πιέζει ο χρόνος και σήμερα περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει αυτή την προσφυγή επί, παραβάση, κατά, επί παραλήψη κατά της Γαλλίας, αλλά να απευθυνθεί και στις ε, ΗΠΑ, ούτως ώστε να γίνει καινούργια επαναδιαπραγμάτευση διεσμερή συμφωνία με τις ε, ευρωπαϊκές Ως και να υπάρξει κάποια εξαίρεση από αυτή την συμφωνία. Ο επόμενος. Ο κύριος Μουσέδα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση. Μου ζητήθηκε να σας μιλήσω 10 λεπτά γιατί ε, ε, ε, προβαίνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επίλυση διαφορών. Για να καταλάβουμε αυτό πρέπει κανείς να εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Η ΦΑΤΚΑ λοιπόν θεσπίστηκε το 2010, προφανώς πρόκειται για έναν εξοεδαφικό νόμο γιατί απαιτεί από ξένα τραπεζικά ιδρύματα να διαβάζουν πληροφορίες στις ΙΠΑ. Οι ΙΠΑ γρήγορα κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη ΦΑΤΚΑ χωρίς τη βοήθεια άλλων χωρών και έγινε προφανές έπειτα από την αναφορά της ΠΕΤΗ, ε, από την έκθεση της ε, ΠΕΤΗ, ότι η κυρία Ιντβελτ βρήκε επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις οποίες και έχουμε εδώ. Το 2011 λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλει επιστολή ε, ε, με ε, θέμα της, τους κατατύχει Αμερικανούς όπου η Κομισιόν δηλώνει ότι υπάρχουν ανησυχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ΦΑΤΚΑ υπάρχουν πιθανές συγκρούσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας με τον, με τον ΦΑΤΚΑ και ότι το, το 2011 όλα αυτά και ότι το κόστος είναι ανησυχητικό. Αυτές, αυτά είναι τα λόγια που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, ξαναλέω, ε, στην επιστολή της. Η δε επιστολή αυτή τελειώνει ε, ε, αναφέροντας ότι ελπίζει ότι μπορεί να θεσπιστεί μια νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να είναι πιο ε, εύκολα εφαρμόσιμη. Άρα από το 2011 η Κομισιόν είναι προφανές ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την εφαρμογή της ΦΑΤΚΑ και την συμβατότητά της με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αν δείτε δε μια άλλη επιστολή την οποία βρήκε η κυρία Ιντβελτ, Μπορώ να προχωρήσω τη διαφάνεια. Ορίστε. Σε ένα επόμενο email της Ταξούντ, ε, δηλαδή της Κομισιόν, σε κατά τύχη Αμερικανό αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Προεδρία και κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διάλογο με τις ΗΠΑ. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούσε γιατί οι ΗΠΑ ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να, να τους διαβιβάσουν πληροφορίες. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει απλώ τι ανησυχίε τη και την ελπίδα τη ότι με τη συνεργασία μα θα μπορέσουμε να καταστήσουμε τον ΦΑΤΚΑ ε, πιο αναλογικό και πρακτικά εφαρμόσιμο. Και εδώ πάλι αναγνωρίζεται από την Κομισιόν ότι δεν είναι αναλογικός ε, ο ΦΑΤΚΑ. Το 2012 η κυρία Ιντφελτ βρήκε μια άλλη ενδιαφέρουσα επιστολή και πάλι τη επίτροπή προς κατατύχη Αμερικανό, όπου αναφέρεται ότι έπειτα από εσωτερική εξέταση σε συνεργασία με τους τη προστασία προσωπικών δεδομένων, η Κομισιόν παραπέμπει το ζήτημα στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που ήταν ε, ο φορέας προστασίας προσωπικών δεδομένων υπό την παλιά οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εκεί αναφέρεται ότι το, η ομάδα εργασίας αυτή ε, επεξεργάζεται μια γνώμη. Αυτά το 2012 με εκείνη την νομοθεσία. Μετά ε, εισέρχεται το ζήτημα αυτό στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τον Απρίλιο του 2012 λοιπόν είχαν γίνει όλα αυτά. Τον Ιούνιο τώρα του 2012, ένα μήνα αργότερα δηλαδή, η ομάδα εργασίας ε, για το άρθρο 29 εξέδωσε γνωμοδότηση για το ζήτημα κατόπιν αιτήματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν δείτε την έκθεση την οποία συνέταξε η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκεί αναφερόταν ότι δεν βλέπει τρόπο να μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ο ΦΑΤΚΑ και τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εξέταση των προσωπικών δεδομένων, αναφερόταν σε εκείνη την γνωμοδότηση, δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Γι' αυτό και θα πρέπει να ξεβρεθούν άλλα μέσα προκειμένου να προστατευτούν και τα δικαιώματα των ε, νομοταγών πολιτών. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση ε, της ΕΠΕΤΗ που εκδόθηκε πέρσι, αναφέρεται ότι κάθε διαδικασία θα πρέπει να σέβεται τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Βάτικα δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε αναλογική. Το 2017 δηλαδή η έκθεση ΠΕΤΗ στην ουσία κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα στο οποίο είχαν καταλήξει η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ήδη από το 2012. Δυστυχώ όμω υπάρχουν πολιτικά ζητήματα τα οποία ε, περιπλέκουν τα πράγματα. Έπειτα από ένα μήνα λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων εξέδωσε εκείνη την καταδικαστική της γνωμοδότηση, ε, οι ΙΠΑ στην ουσία ε, προχώρησαν στην έκδοση του, πρώτη, του, του προτύπου για τις διακυβερνητικές συμφωνίες που θέλουν να συνάψουν με τα κράτη-μέλη. Διμερός. Εκείνοι λοιπόν εξέδωσαν αυτέ τι συμφωνίε που του επέτρεψαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν τι σχετικέ πληροφορίε που χρειάζονται υπό τον ΦΑΤΚΑ. Μέσα σε δύο μήνε λοιπόν, οι πρώτε χώρε, τα πρώτα κράτη-μέλη, άρχισαν να συνάπτουν τέτοιες συμβάσει με τις ΗΠΑ και το έκαναν αγνοώντας τις ανησυχίες της Κομισιόν, αγνοώντας τις συμβουλές, τις νομικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το έπραξαν αυτό διότι πολλές ε, ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν προβλήματα με τις ΗΠΑ που τους είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ ε, πρόστιμα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και γι' αυτό έπρεπε να βρεθεί γρήγορα μια λύση. Υπήρξε λοιπόν μια μεταστροφή εδώ. Θυμάστε το πρώτο email όπου η Κομισιόν εκφράζει τις ανησυχίες της για τον ε, ΦΑΤΚΑ. Τι έγινε μετά. Δεν ξέρω αν έγινε εδώ, αλλά πέρσι έγινε μια ακρόαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε ότι δεν είναι ρόλος του Συμβουλίου να αξιολογεί τις επιπτώσεις διακυβερνητικών συμφωνίων, συμφωνιών που συνάπτουν τα κράτη-μέλη, διότι είναι διμερείς συμφωνίες. Το 2011 όμως το Συμβούλιο βρισκόταν σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τώρα πια λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με εμά αυτό το θέμα. Ε, αυτό είναι ε, προσβλητικό για τους ε, νομοταγείς πολίτες. Ακόμη και η Επίτροπος ε, είπε ότι σας ευχαριστώ που μας ε, ε, θέτετε και που εφιστάτε την προσοχή μας σε αυτά τα ζητήματα. Μα τα ζητήματα αυτά είναι γνωστά εδώ και 9 χρόνια. Τα φορολογικά ζητήματα ε, υποτίθεται ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Μα αυτό δεν ισχύει διότι ήδη από το 2011 ε, το ζήτημα δεν ε, περιορίζεται σε φορολογικά θέματα, αλλά αφορά και την προστασία δεδομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ουσία. Πρόκειται για ανταλλαγή πληροφοριών στη βάση αμερικανικών κριτηρίων για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Στην ουσία πρόκειται για μια ε, επίφαση διαφάνειας η οποία καταστρατηγεί κάθε έννοια ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητα πληροφοριών. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, μια σειρά από ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εθελοτυφλούν Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που διαδέχθηκε την ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Γνωρίζουμε και από τον τύπο ότι ο ΦΑΤΚΑ Νόμιζα ότι είχα άλλα 40 δευτερόλεπτα, λέει ο μιλητή. Τέλο πάντων, εντάξει. Ε, υπήρξε νομική προσφυγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ε, έχει εισόδημα κάτω από 140 δολάρια το χρόνο ε, και ε, ως εκ τούτου δεν, δεν είναι φόρου στις ΗΠΑ Τη ζητήθηκε πάντως παρόλα αυτά να ε, κοινοποιήσει τις, ε, τα προσωπικά της δεδομένα. Ε, την προηγούμενη, πέρσι η Washington Post εξέδωσε άρθρο στο οποίο κατακρίνεται σφόδρα το μηχανογραφικό σύστημα των, που χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές, διότι είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει από το 1960, από τη δεκαετία του 1960 και σε κάθε περίπτωση παραβιάζεται ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε ο καθένας 10 λεπτά. Αλλά επειδή στις 12.30 θα σταματήσει η διερμηνία, είπαμε ότι έχει 8 λεπτά ε, ο κάθε ομιλητή μας. Κυρία Λίσσα Μπέικιμαν. Βέικιμαν, συγγνώμη, είναι η επόμενη. Έχετε και εσείς 8 λεπτά από τη Γενική Διεύθυνση Just της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ε, θα μιλήσω για τους κανόνες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν ε, θα αναφερθώ στον ε, χειρισμό των δεδομένων στο πλαίσιο του ΑΦΚΑ και τι ε, διασφαλίσεις που υπάρχουν στο τομέα αυτών. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα αναθεώρησε τους κανόνες της για προστασία των δεδομένων και ε, η σχετική νομοθεσία ε, τέθηκε σε ισχύ πέρσι. Ε, η νομοθεσία αυτή αντικατέστησε την προηγούμενη νομοθεσία που ίσχυε επί πάνω από 20 χρόνια. Το GDPR έχει επικαιροποιήσει τους κανόνες, δεν έχει όμως αλλάξει ριζικά αυτό που ίσχυε πριν. Το ο κανονισμό λοιπόν για την προστασία των δεδομένων ε, θεσπίζει τι ε, βασικέ αρχέ ε, για όσου χειρίζονται προσωπικά δεδομένα και αυτό ισχύει και για ιδιωτικού φορεί και για αρχέ. Υπάρχει λοιπόν η αρχή του περιορισμού του στόχου. Διακόπτη η πρόεδρο. Παρακαλούμε λίγο πιο αργά. Και ε, δίνει κάτι, ε, κάποια δικαιώματα σε ιδιώτες, για παράδειγμα την πρόσβαση στα δεδομένα του καθενός ή να πετύχει ε, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι ότι ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων θεσπίζει και κανόνες για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες ή άλλους οργανισμούς. Όταν αποστέλλονται δεδομένα σε τρίτη χώρα, οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τις διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων. Όλοι οι φορείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται στον GDPR και ε, όταν χειρίζονται δεδομένα στο πλαίσιο του ΦΑΤΚΑ. Συγκεκριμένα λοιπόν όσον αφορά τις διασφαλίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο του ΦΑΤΚΑ. Παρέχονται μέσα από ένα συνδυασμό διαφόρων ε, μέσων, διεθνών ε, συμφωνιών, ε, διοικητικών ρυθμίσεων ε, και άλλων ε, διεθνών μέσων στον τομέα της συνεργασίας πάνω σε φορολογικές υποθέσεις. Όπως τόνισαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ε, ο ΦΑΤΚΑ εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη μέσω ε, διακρατικών ε, συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί παραπέμπουν στην επιστευτικότητα και προστασία που παρέχεται σε άλλες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείε και τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ή του ΟΣΑ για την διοικητική συνεργασία σε φορολογικές υποθέσεις. Η σύμβαση αυτή και άλλες ε, διακρατικέ ε, συμφωνίε, άλλες διμερεί ε, συμφωνίε περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίε που ανταλλάσσονται με τι ΗΠΑ. Οι πληροφορίε αυτές ανταλλάσσονται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και σχετικό. Και τέλος, η σύμβαση αυτή Λέει επίσης ότι τίποτα εντός της ε, συμφωνίας ε, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που παρέχονται σε άτομα μέσω του διεθνούς δικαίου. Και οι κρατικές αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης επόκεινται απολύτω στον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να, να συμμορφώνονται με τις αρχές για την προστασία των δεδομένων, να διασφαλίζουν την διαφάνεια και να επιτρέπουν ε, στα άτομα συμπεριλαμβανομένων αυτών με διπλή υπηκότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους. Επιπλέον ε, υπάρχει η Εθνική Νομοθεσία που εφαρμόζει τις ε, διεθνείς συμφωνίες οι οποίες μπορεί να καθορίζουν περαιτέρω τις υποχρεώσεις φορέων στο πλαίσιο του ΦΑΤΚΑ. Πολύ συγκεκριμένες διατάξεις για την διαφάνεια απέναντι σε άτομα, για παράδειγμα, ή το διάστημα διατήρησης των δεδομένων. Επιπλέον, ε, όλοι οι μηχανισμοί προσφυγής ε, στο πλαίσιο του ε, κανονισμού για την προστασία των δεδομένων είναι διαθέσιμοι σε όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν λοιπόν να ζητήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων τους και μπορούν να ε, προσφύγουν και στα εθνικά δικαστήρια στα κράτη-μέλη. Από ό,τι γνωρίζουμε, μέχρι στιγμή ε, δεν έχουν υπάρξει προσφυγή ε, στι αρχές προστασίας δεδομένων της ευρωπαϊκή Ένωσης. Τούτου λεχθέντος, οι αρχές προστασίας δεδομένων εξέτασαν το θέμα αυτό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν περιπτώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή όπου έπρεπε να παρέμβουν. Βέβαια ε, υπάρχουν και ανεξάρτητοι ε, φορείς εφαρμογής ε, των κανόνων προστασίας δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και αυτοί είναι πιο κατάλληλοι να εξετάσουν το θέμα αυτό. Επίσης έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, όπου συγκεντρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι φορείς προστασίας δεδομένων των κρατών μελών. Παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις εκεί πέρα. Μέχρι στιγμή, από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχουν υπάρξει προσφυγές σε εθνικές αρχέ προστασία δεδομένων, έχουν υπάρξει δικαστικές υποθέσεις ε, και ε, όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις ε, στα κράτη-μέλη. Ε, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδικίες που ήδη υπήρξαν, θα ήθελα να τονίσω ότι το υψηλότερο δικαστήριο τη Γαλλία, το Conseil d'État, εξέτασε ε, συγκεκριμένα την ε, Γαλλική ε, Συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε για το ΦΑΤΚΑ και διαπίστωσαν ότι δεν παραβιάζει ούτε τα θεμελιώδη δικαιώματα ούτε την προστασία δεδομένων. Μάλιστα, σημειώνει ότι και η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών παρέχει κάποιες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων στον τομέα αυτών. Για παράδειγμα, την δυνατότητα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων των, των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα προσφυγής ε, στα Αμερικανικά δικαστήρια για τέτοια θέματα. Υπό το φως όλων αυτών των εξελίξεων, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και ε, την συγκεκριμένη προσφυγή, η οποία έχει υποβληθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όσον αφορά την Γαλλική Συμφωνία. Την λάβαμε πριν κάποιες εβδομάδες ε, και ε, επιβεβαιώσαμε απέναντι στον Τούντα ότι έχει καταγραφεί και εξετάζεται η προσφυγή του και θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο μιλήτρη, αν μίλησα πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον τήρησα το χρόνο ομιλίας μου. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρία Λίσσα, <laughs> Α, όχι. Έκανα λάθος, έκανα λάθος. Η κυρία Ισμήνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα ξεκινήσω πρώτα παρουσιάζοντας ε, το έργο ε, του επόπτη και του προκατόχου του, της ομάδας εργασίας για το άρθρο 29 σχετικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, ιδίως με έμφαση στο ΦΑΤΚΑ και από εκεί και πέρα θα μιλήσω και λίγο για τη δουλειά που κάνει ο EDPB για το ζήτημα αυτό. Ο EDPB και η ομάδα εργασίας για το άρθρο 29 έλαβαν μια σειρά αποδράσεις όσον αφορά τον ΦΑΤΚΑ και την αυτόματη αυτόματη ανταλλαγή προσωπικών φορολογικών δεδομένων τα τελευταία 7 χρόνια. Ο EDPB και η ομάδα εργασίας έχει εκδώσει από το 2012 έξι έγγραφα ε, συμπεριλαμβανομένων επιστολών, δηλώσεων και κατευθυντηρίων γραμμών. Να ξεκινήσω με τις επιστολές του 2012 που συνέταξε η ομάδα εργασίας ε, του άρθρου 29 στην ε, φορολογική μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί τονίζεται η ανάγκη να υπάρχει νομική βάση για ε, την νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ΦΑΤΚΑ. Τονίσαμε ότι η απουσία τέτοιας νομικής βάσης μπορεί να οδηγήσει σε εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων στην απαγόρευση της διαβίβασης ε, προσωπικών δεδομένων, καθώς κάτι τέτοιο θα, θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της εθνικής νομικής ε, ε, νομοθεσίας μάλλον για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα υποστηρίζαμε ότι κάθε διαβίβαση πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται με ταυτόχρονο σεβασμό στους κανόνες προστασίας δεδομένων. Είπαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει με νομικά δεσμευτική συμφωνία για παράδειγμα χρησιμοποίησαμε την, την ε, αρχή της αναλογικότητας είπαμε ότι θα πρέπει να το, τονίζεται η να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων των δεδομένων και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων. Με βάση λοιπόν τις συστάσεις της ομάδας εργασίας του 2012, τα κράτη-μέλη άρχισαν να υπογράφουν διακυβερνητικές συμφωνίες με την Αμερικανική κυβέρνηση, δημιουργώντας στην ουσία αυτή τη νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του ΦΑΤΚΑ. Οι περισσότερες από αυτές τις ε, συμφωνίε συμφωνίες υπογράφηκαν μεταξύ 2013 και 2016. Το 2015 η ομάδα εργασία εξέδωσε νέα δήλωση και μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές ε, όπου υπενθύμιζε τις αρχές ε, και τις διασφαλίσει προστασία προσωπικών δεδομένων που πρέπει να γίνονται σεβαστές στις ε, διακρατικές ανταλλαγέ προσωπικών δεδομένων για φορολογικού σκοπού. Αυτό έγινε προκειμένου να ε, ε, ε, υπενθυμιστεί στις κυβερνήσεις ότι πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι, τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και ιδίως η αναλογικότητα και η αναγκαιότητα. Το 2018 η ομάδα εργασίας 29, του άρθρου 29 απάντησε σε αιτήματα της Ένωσης κατά των κατατύχη Αμερικανών να ε, δώσει τις δικές της απόψεις σχετικά με το ΦΑΤΚΑ και ιδίως τη θέση της για τους ε, κατατύχει Αμερικανούς. Σε αυτά τα αιτήματα η ομάδα εργασίας ε, απάντησε υπενθυμίζοντας καταρχάς τις δράσεις που είχαν αναλυφθεί μεταξύ 2012 και 2018. Επίσης τονίσαμε ότι ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει περίπτωση όπου η Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων χρειάστηκε να απαγορεύσει την διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών υπό το καθεστώς του ΦΑΤΚΑ. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του ΦΑΤΚΑ, η ομάδα εργασίας τόνισε ότι δεν είναι αρμόδια να απαντήσει και το ίδιο ισχύει και σήμερα για τον EDPB. Η ομάδα εργασίας υπενθύμησε τις εναλλακτικές που έχουν στη διάθεσή τους οι κατατύχει Αμερικανοί και όποιος άλλος έχει επηρεαστεί αρνητικά από τον ΦΑΤΚΑ. Μπορούν να απευθύνονται σε εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. Υπάρχουν και άλλες νομικές οδοί, όπως για παράδειγμα ε, η προσφυγή σε εθνικά δικαστήρια, την οποία επίσης έχει αξιοποιήσει η Ένωση κατά τύχη Αμερικανών με την προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας. Επίσης, καμία εθνική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν έχει λάβει καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πολιτών στο πλαίσιο της ΦΑΤΚΑ, ούτε και στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών που έχουν υπογράψει οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ. Για την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν μπορεί να ε, εγκρίνει ε, δεν έχει ακόμη, αλλά μάλλον εργάζεται επί της, για την επεξεργασία συγκεκριμένων κατευθυντήνων γραμμών ε, για, τις ευρωπαϊκές, για τις εθνικές αρχές ε, προστασίας δεδομένων. Δεν απαντούμε δηλαδή σε μεμονωμένα εξατομικευμένα αιτήματα πολιτών, αλλά προσπαθούμε ε, και θα ολοκληρώσουμε ε, στο προσεχές διάστημα την σύνταξη των καθηγητήριων γραμμών για τα άρθρα 46.2 και 46.3 του GDPR. Πιο συγκεκριμένα, το EDPB προσπαθεί με αυτές τις κατευθύνες γραμμές να δώσει συγκεκριμένες και χρήσιμες ε, οδηγίες για την προετοιμασία και τη σύναψη νομικά δεσμευτικών και εφαρμοστέων μέσων που θα έχουν υπογραφεί μεταξύ δημοσίων αρχών ή κρατικών φορέων. Αυτά, αυτές οι κατευθύνες γραμμές θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κράτη-μέλη και τις εθνικές αρχές ε, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις ε, διακυβερνητικές συμφωνίες και με την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε τροποποίηση των διακυβερνητικών συμφωνιών και την ευθυγράμμιση αυτών με τις απαιτήσει του GDPR. Ελπίζουμε ε, να ολοκληρώσουμε την σύνταξη αυτών των καθημερινών γραμμών εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για 6 έως 8 εβδομάδες πριν από την τελική τους ε, έγκριση αμέσως μετά την περίοδο διαβούλευσης. Πάρα πολύ και τώρα να δώσουμε στα μέλη της Επιτροπής το λόγο. Κάποιος συνάδελφος θέλει να λάβει το λόγο. Κυρία Κερδοντάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι μερικές φορές όλη αυτή η συζήτηση για, τη, για την ΦΑΤΚΑ φαίνεται καυκακική. Και το βάρος πέφτει στους ώμους του ατόμου που πρέπει να βρει τρόπο να βγει από το λαβύρινθο του νομικού πλαισίου και των διαφορετικών νομοθεσιών, είτε πρόκειται για την προστασία δεδομένων, ε, τον τραπεζικό τομέα ή τις διακρατικές συμφωνίες. Ανά πάσα στιγμή ε, τους λέμε ότι μπορούν να προσφύγουν, ε, υπάρχουν ένομα μέσα. Αλλά απαιτεί πολύ μεγάλους πόρους από το πρόσωπο να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους ε, και Φαίνεται στη συζήτηση αυτή να μην ε, λαμβάνεται υπόψη καθόλου αυτός ο παράγοντας. Η ερώτησή μου είναι, μήπως ως αποτέλεσμα των ε, διμερών ε, συμφωνιών και συμπεραίνοντας από την προηγούμενη παρέμβαση ότι υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες που πρέπει να αναθεωρηθούν ως αποτέλεσμα των κατευθυντηρίων γραμμών Υπάρχει λοιπόν μια... Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των κατά Αμερικανών σε, διάφορα, σε, σε κάθε κράτος μέλος. Διαφέρει λοιπόν η νομοθεσία αρκετά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Σε τι βαθμό αυτό προκαλεί ανησυχία στις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων που επιθυμούν εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και θίγω το θέμα αυτό, διότι συμπεραίνω από τις ε, επίσημες παρεμβάσεις ε, σχετικά με το τι έχει σχεδιαστεί, ότι έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να συγχαρώ το συνάδελφο που αποκάλυψε όλα τα ε, έγγραφα που έχει αποκαλύψει η αυτά τα τελευταία χρόνια. Μήπω, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων ε, έχουμε μία λοταρία αναταχυδρομικό κώδικα, δηλαδή ότι, ε, ότι διαφέρουν οι κανόνε ανάλογα με το που βρίσκεται κανεί. Ευχαριστώ πολύ, ο Πίτερ. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό και έτσι μπορούμε σιγά σιγά να φτάσουμε στα σημερινά μα συμπεράσματα. Διότι έχω καταγράψει εδώ πέρα. Φανταστείτε να έχετε μια ε, υπηκότητα την οποία δεν επιθυμείτε καθόλου και δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε το αρχικό λάθος που έχει να κάνει με το ότι στον φορολογικό τομέα το κάθε κράτος μέλος αποφασίζει μόνο του και έτσι πρέπει να προσφύγει σε διμερείς συμφωνίες. Ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, διότι μέχρι τώρα λέει ότι δεν μας αφορά καθόλου. Είναι λάθος αυτό, δεν επιτρέπεται να το, να το αφήσουμε αυτό να περάσει, διότι έχει να κάνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, πολιτών και έχει να κάνει με την προστασία των δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση. Άλλωστε έχουμε τελείω άλλο ε, ειδικό βάρο εάν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει στο όνομα όλων των φορέων. Και ε, εάν συνεχίσουμε τις διακρατικές συμφωνίες, τότε έχουμε μια ακόμη πιο παρανοϊκή κατάσταση, διότι θα εξαρτάται η κατάσταση του καθενός από το που διαμένει, αν μένει στη Γερμανία, στην Ελλάδα κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι οι πολίτες αυτοί είναι δικοί μας ε, υπήκοοι και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιμπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και πάλι τους ομιλητές. Να πω και πάλι στον κύριο Νοσέδα ότι πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα έγγραφα που καταφέραμε να αποκαλύψουμε. Δύο ρητορικά θα πω ε, ερωτήματα προς την Κομισιόν. Γιατί νομικά ένδικα μέσα μιλάτε ακριβώς. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι κάποιος που βρίσκεται στην Ευρώπη αποκλείεται ή δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικές πληροφορίες, ε, υπηρεσίες στην Ευρώπη. Και εσείς μιλάτε για ένδικα μέσα στη ΣΥΠΑ. Για ποιο ακριβώς αντικείμενο. Ανοησίες. Δεύτερον, η Κομισιόν επιμένει πάντοτε ότι πρόκειται για φορολογικό ζήτημα και αυτό αυτόν τον λόγο μπορεί να επιληθεί μόνο μέσω διμερών συμφωνιών, καθώς η φορολογία είναι εθνική αρμοδιότητα. Ανοησίες και πάλι. Δεν πρόκειται για φορολογικό ζήτημα. Η IGA συνήθισαν για συμμόρφωση με, ευρωπαϊ... με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, που είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, ενωσιακή αρμοδιότητα. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο η Κομισιόν μπορεί να προτείνει Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση είπα, για την υπεράσπιση και την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Καμία σχέση με φορολογία. Φαντάζομαι βεβαίω ότι δεν μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Απλώ διαβιβάστε το στους ε, πολιτικά ανωτέρους σας, τους ε, πολιτικά υπεύθυνους ε, επιτρόπους και εκείνους που θα αναλάβουν σύντομα τα καθήκοντά τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία... Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Βάκεμαν, γιατί εκείνη αφορούσαν λύσω τα περισσότερα ερωτήματα. Ευχαριστώ για τον πιθανό κίνδυνο διαφορετικών προσεγγίσεων στα κράτη-μέλη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε και κατά την συζήτηση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Ως προς αυτό θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενδείξεις ότι θα υπάρχει διαφορά στο πώς ε, θα, τι, τι, ε, σε τι επεξεργασία θα τεθούν τα δεδομένα μεμονωμένων ατόμων, διότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν συνάψει την ίδια στην ουσία διακρατική συμφωνία διμερός με τις ΗΠΑ καθώς και τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΣΑ που, έχει, που περιλαμβάνει τις παρόμοιες ε, εγγύησεις. Όσον αφορά την προστασία δεδομένων, ο GDPR ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης, οπότε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία ότι μπορεί να εμφανιστεί μια τέτοια διαφορετική προσέγγιση. Όταν συνήθισαν αυτές οι, οι διεθνείς συμφωνίες, οι διακρατικές, δια, διακυβερνητικές συμφωνίες, συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή και πάρα πολλέ εθνικές ε, αρχές προστασίας δεδομένων και τι ενέκριναν και όπω είπα πέρσι σε, σε ενωσιακό επίπεδο οι εθνικέ αρχέ ε, προστασία προσωπικών δεδομένων ε, δημοσίως δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις όπου παραβιάστηκαν οι κανόνες προστασίας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και για να επανέλθω και στα ζητήματα που τέθηκαν σε σχέση με τα ένδικα μέσα που ανέφερα. Η παρουσίασή μου βεβαίως αφορούσε την διάσταση της προστασίας των δεδομένων. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι μιλούσα για τα ένδικα μέσα που ε, προβλέπονται από το GDPR στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπε και στην απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας, Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, υπάρχει νομοθεσία ε, η οποία διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω ε, από μάλλον δημόσιους φορείς και σε, αυτούς, σε αυτή την νομοθεσία ε, περιλαμβάνονται και στα ένδικα μέσα που προσφέρονται περιλαμβάνονται και τα ένδικα μέσα για την προσφυγή σε αμερικανικά δικαστήρια. Για την φορολογία, ε, για το αν το ζήτημα αφορά τη φορολογία ή την προσωπικά δεδομένα, εγώ δεν θα απαντήσω. Θα αφήσω σε αυτό το ερώτημα να απαντήσουν οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος Κομισιόν που θα ήθελε να τοποθετηθεί. τελειώνουμε αυτό το σημείο της ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, αναφέροντα και όσου έλαβαν τον λόγο αλλά και τους προσκεκλημένους μας. Αλλά θέλω να σας πω το πιο σημαντικό, ότι από πλευρά της Επιτροπής μας, ότι όλες, όλες οι πολιτικές ομάδες, όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου συμφωνώ θα πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, συμπολίτες μας για αυτό το θέμα. Όχι, αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα. Δεν θα τους εγκαταλείψουμε. Η Επιτροπή των Αναφορών είναι η πύλη, η πύλη η επικοινωνία, η γέφυρα των πολιτών με τα θεσμικά όργανα και όχι μόνο με το Κοινοβούλιο. Οπότε, ω Επιτροπή Αναφορών, θα απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε ουσιαστικά να προσπαθήσει να βρει μια ε, λύση, να υποστηρίξουμε του ε, πολίτε, ε, γιατί ακριβώ αυτό θέλει να ζητήσει η Επιτροπή μας. Και ολοκληρώσαμε την πρωινή συζήτηση, είχαμε ένα σωρό προτάσεις, οπότε θα ζητήσουμε να βρει λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ το λόγο κυρία Ενετφέλντ. Πέραν αυτού... Μπορείτε επίσης παρακαλώ να ε, ακολουθήσετε την πρότασή μου να στείλετε επιστολή στην ε, Φιλανδική Προεδρία. Ναι, φυσικά και μόλις έχουμε τους ε, νέους επιτρόπους. Επιτροπός μας ε, θα είναι ο Αντιπρόεδρος ε, κύριος Σεύκοβιτς. Υποσχέθηκε να επισκέφτεται την Επιτροπή μας σε τακτική βάση κάθε εξάμεινο ή κάθε χρόνο. θα τα διαβάσουμε αυτά στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Νετφέλτ, ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Φιλανδική Προεδρία, ε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε, πρέπει να του στείλουμε επιστολή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Άλλωστε, οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι προσπαθούν να πετύχουν ε, οι Φιλανδοί να αναλάβουν πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν θα το κάνουμε αυτό. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ όλους. Λήξη της ακρόασης.